Γέννη ζώφτης. Οι συντάκτες. Η κυρία Χάουτελα, δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την προηγούμενη συζήτηση και να πω ότι όντω είμαι η πρόεδρο τη Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και έστειλα μια επιστολή στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου όπου ζητούσα να ε, προωθηθούν οι συζητήσεις αυτές ούτως ώστε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμμετάσχουν με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη τους σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί το κύρος του Κοινοβουλίου υπονομεύεται πάντοτε από την τόσο μικρή παρουσία μας εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το Καζακστάν είναι μια σημαντική χώρα στην Κεντρική Ασία και θα αναλάβει του χρόνου την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε ούτως ώστε να τιμωρούνται ε, με τον ε, κατάλληλο τρόπο τα εγκλήματα σε μια χώρα που θα αναλάβει τόσο υψηλά καθήκοντα του χρόνου. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση του Γευγένη Βόφτης, ο οποίος ε, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξαμελίας και καταδικάστηκε σε τετραετή κάθυρξη αφού χτύπησε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν πεζό. Λαμβάνοντας επίσης ε, υπόψη το γεγονός ότι και στον ίδιο τον ΟΑΣΕ ε, ακούστηκαν ε, ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον παραβιάστηκαν οι αρχές μιας δίκαιης δίκης. Αυτό είναι μια αρχή που εγγυάται το Σύνταγμα του Καζακστάν συζητήσαμε το θέμα αυτό και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, ούτω ώστε να πιέσουν και αυτοί από την πλευρά τους για μια δίκαιη δίκη. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει λόγο ε, για το πώς οι χώρες της Κεντρικής Ασίας ενισχύουν ε, την αρχή του κράτους δικαίου και αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παλακής έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΣΕ. Ε, Παρ' αυτά, ε, το Καζακστάν ε, απέχει πολύ από τα διεθνή στάνταρ, τα διεθνή πρότυπα. Είναι μια χώρα που δεν ακολουθεί τις συστάσεις του ΑΣΕ. Ε, Πραγματικά υπάρχουν πολλές παραβιάσεις ε, του νόμου και των θεμελιδών αρχών και ε, δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτή η χώρα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, παραβιάζεται η ελευθερία του τύπου και πολλές άλλες αρχές. Στην περίπτωση του Σβαγένη Σβόφτιτς του Ραμαζάν Γεσέρκοφ και του Σεργέη Ντουβάνοφ ε, καλούμε το Καζακστάν να ε, σεβαστεί ε, τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι δίκες πρέπει να, είναι, να με αμερόληπτο τρόπο και αυτοί που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να υφίσταται τέτοιες συνέπειες στην επόμενη φάση του ε, διαλόγου με το Καζακστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Οκτώβριο ε, θα θέλαμε να καλέσουμε το Συμβουλίο να ε, θέσει τα ζητήματα αυτά και η Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί ώστε η ανάληψη των καθηκόντων από το Καζακστάν του χρόνου να μην υπονομεύσει όλα, όλες αυτές τις αρχές. Would like to express my sympathy to the... Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τη συλληπιτήριά μου για το τροχαίο ατυχήμα στο οποίο έχασε τη ζωή του κύριου ε, ε, Ζόβτης. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου για την κατάσταση ε, του κυρίου Ευγένη Ζόφτης. θα πρέπει όλοι να δειχθούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται κυρώσεις. Και ο κύριος Ζόφτης ε, είναι ένας ε, δικηγόρος, αν και μετά που το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη. Ο κύριος Ζόφτης δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί για οτιδήποτε άλλο από το τροχιό ατύχημα στο οποίο είναι πλάκια. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τιμωρηθεί για τις δραστηριότητες του ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επειδή ήταν κρίσιμη και κριτική φωνή στο Καζακστάν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό οι δικαστικές αρχές του Καζακστάν να διεξάγουν ε, έρευνες με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου, να υπάρχει υπάρχει μια σωστή και δίκαιη έρευνα στις συνθήκες που οδήγησαν στο ε, τύχημα αυτό και να αναθεωρήσουν την καταδίκη ε, και την έκτηση ποινής εκ μέρους του κυρίου Ζόφτης. Τον λόγο έχει η κυρία Γίγκλε. Ε, πρόεδρε, αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα εξεπλάγει λιγάκι για τη νομική αξιολόγηση ενός ε, τραγικού τροχαίου ατυχήματος, ένας μοιραίου, ε, γιατί θεώρησε ότι αυτό αιτιολογεί το να μπει το θέμα ως θέμα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μας είναι σημαντικό το ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από έναν εξάρτητο δικαστήριο καταρχήν δεν αμφισβητούνται, εκτός βέβαια αν πρόκειται για ε, δίκες μαριονέτες, ε, κάτι που ζήσαμε παραδείγματος χάνη, στο Ιράν. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Για μας ε, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι η πεμπτουσία της ε, δημοκρατικής τάξης πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν την απόφαση αυτή καταρχήν πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Κατόπιν θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι ένας άνθρωπος ε, βέβαια έχασε τη ζωή του σε αυτό το τροχαίο τύχημα. Γι' αυτό λυπούμεθα, εκφράζουμε τη λύπη μας, όμως ε, έλαβε χώρα και νομική και δικαστική έρευνα. Το γεγονός ότι ο κύριος Οφτής εμπλέκεται στο θέμα αυτό ε, που είναι υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό τράβηξε την προσοχή επάνω του και οδηγεί στο να ασχολούμαστε και εμείς με αυτή την υπόθεση σήμερα. Το ΕΛΚ αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Καζακστάν να επιτύχει πρόοδο στον δρόμο της δημοκρατίας και της ε, ευνομίας και διαβεβαιώνει το Καζακστάν για την αμέριστη υποστήριξή του. Ενθαρρύνει το Καζακστάν να συνεχίσει αυτή την πορεία με ε, κατηγορηματικό και αποφασιστικό τρόπο. Καλούμε τις αρχές του Καζακστάν ε, προς ίδιον να δώσουν εκτενείς πληροφορίες ε, στη δημοσιότητα, να παρουσιάσουν την δική τους ε, την άποψη και στον κύριο Σβώτης να διασφαλίσουν μια δίκαιη ε, διαδικασία κατάθεση εφέσεων. Το Καζακστάν εδώ αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον, ένα λεπτό. Πρόεδρε, συμφωνώ με την κυρία Γέγκλε. Πραγματικά είμαι αποσβολωμένος που ολόκληρο το Στρασβούργο εδώ ήρθε να συζητήσει στα κατεπίγωνα για ένα τροχαίο στο Καζακστάν, στο οποίο σκοτώθηκε τραγικά ένα άτομο και ο οδηγό του αυτοκινήτου τυχαίνει να είναι ένα αγωνιστή των δικαιωμάτων του, του ανθρώπου και από δικαστήριο νόμιμα καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση. Σε και ότι αυτή η φυλακή χαμηλής ασφάλειας έγινε κατα... στρατόπεδο κατα... ποινικό στρατόπεδο στο κείμενο του ψηφίσματος. Πραγματικά είναι κάτι που μειώνει την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Εμείς ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποδυναμώνεται, υποτιμάται όταν αρχίζουμε να συζητάμε για το Μα λέμε ότι η κυβέρνηση του Καζακστάν πέταξε κάτω από τους τροχούς του αυτοκινήτου ενός αγωνιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έναν πολίτη. Λέμε ότι ε, η ποινή Ενό ανθρώπου που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξαμελία είναι πολύ μεγάλη. Ε, δεν μπορούμε να, συνεχίζουμε να καταδικάζουμε το Καζακστάν για πολιτικού λόγου, προσπαθώντα να μειώσουμε ε, την αξιοπιστία ε, της επόμενης προεδρίας του ΑΣΕ. Πραγματικά κάτι τέτοιο είναι, είναι ντροπή που είναι στην ημερήσια διάταξη αυτό το κείμενο και ελπίζω να υποστηριχθούν τροπολογίε από του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το, κύριο λόγο, το λόγο έχει ο κύριο ε, Κολτσεφτσόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω παρόμοιες αμφιβολίες κι εγώ, όπως και ο κύριος Στίβενσον. Το Καζαχστάν είναι μια σημαντική χώρα, όντως. Κάνει τεράστιες προσπάθειες στο δρόμο προς τη δημοκρατία. Δεν είναι πραγματικά ακριβώς ένα υπόδειγμα ε, δημοκρατίας, αλλά επειδή την ξέρω αρκετά αυτή τη χώρα, μπορώ να πω ότι η κατάσταση τώρα στο Καζακστάν είναι πολύ καλύτερη από ότι σε μια σειρά από γειτονικέ του χώρες στην ίδια περιοχή. Ευτυχώ δεν έχουν τέτοια προβλήματα ε, σαν αυτά που υπάρχουν στη Ρωσία που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και συμφωνώ με τον κύριο Στέβενσον ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ρίχνει το κύρος του ε, για το θέμα μιας ε, απλής δικαστικής υπόθεσης. Κάποιες εξηγήσεις πρέπει να δοθούν εδώ, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ε, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε ε, αυτό το ψήφισμα. Αποδυναμώνουμε τη φωνή του Κοινοβουλίου όταν ε, το Κοινοβούλιο αρχίζει να ζητάει θέματα που δεν αξίζουν την προσοχή του. Oh, catch the eye. Ξεκινάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Καζαχστάν ε, διαδραματίζει σημαντικό ε, οικονομικό ρόλο και ρόλο ασφάλειας στον κόσμο. Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, βελτιωθεί. Πέρυσι μάλιστα ακούσαμε εδώ τον πρόεδρο του Καζακστάν. Παρά τον ε, διεθνή έλεγχο ε, δυστυχώς ε, υπάρχει μεγαλύτερη λογοκρισία στη χώρα και λιγότερη ελευθεροτυπία. Βλέπουμε ότι συλλαμβάνονται όλο και περισσότεροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ο κύριος Ευγέννη Ζόφτης, αγωνιστής, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Και νομίζω ότι αυτό ε, βάζει ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο είναι ικανό το Καζακστάν να λάβει την Προεδρία στον ΟΑΣΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόσελτε, πρόεδρε, καταρχήν θέλω να σας πω χαίρομαι που είναι πίσω η Χάιντι Χάουταλα, αλλά για κάποια χρόνια έλειψε από εδώ. Και ξέρετε ε, τότε υπήρχε εδώ το Συμβούλιο την Πέμπτη το απόγευμα. Η Τσεχική και η Γερμανική Προεδρία ήταν παρούσες εδώ την Πέμπτη το απόγευμα. Και εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναβάλουμε τις συζητήσεις. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα την Τετάρτη το απόγευμα. Πρέπει να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να είναι παρόν την Πέμπτη εβδομάδα και να μην συζητιούνται όλα τα θέματα την Τετάρτη. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, πράγματι, εδώ πιστεύω ότι πρόκειται μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά ακριβώ γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Καζακστάν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να επιμείνουμε στο να υπάρξει αντικειμενική έρευνα. Εδώ λοιπόν υποστηρίζω απόλυτα την κυρία Γίγκλε. Για τον λόγο αυτό υπογράψαμε το ψήφισμα. Πρέπει να υπάρξει ε, μια απόλυτα αμερόληπτη έρευνα για το θέμα αυτό που δεν θα συγκαλύπτει απολύτως τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που λάβατε το λόγο και θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο στην Επίτροπο. Με μεγάλη ανησυχία σημειώσαμε τα θέματα αυτά των ε, ε, ομών παραβιάσεων ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως όσον αφορά τον κύριο Ζόφτης, ο οποίος καταδικάστηκε για δολοφονία μετά από αυτό το μοιραίο τροχαίο ατύχημα. Όπως ξέρετε, οι αρχές του Καζακτάν απέρριψαν το ότι υπήρχαν πολιτικά κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η Κομισιόν στηρίζει απόλυτα το, τη δήλωση της ε, Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της 10 Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ ε, σοβαρό το θέμα και πρέπει να υπάρξει μια πολύ προσεκτική και δικημενική έρευνα. Κανούμε λοιπόν το Καζακστάν που είναι η επόμενη χώρα πρόεδρος ε, στο, ε, στον ΟΑΣΕ να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ε, Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί το όλο θέμα εκ του σύνεγγης. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Τώρα θα συζητήσουμε έξι σχέδια ψηφίσματος για την Συρία, ιδίως δε την υπόθεση του μοναδ Αρχασανή. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. Η κυρία Φρανσίσκα Μπράτνερ, δύο λεπτά.